Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε ενσωμάτωση των δύο συστημάτων. Και γιατί θα έπρεπε, γιατί να μην υπάρχει ένας ανταγωνισμός ανά την Ευρώπη, να έχουμε, γιατί να έχουμε ένα μονοσύλλαβο σοβιετικό σύστημα που το αποφασίζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Επιτροπή, δεν θα λειτουργήσει. Πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός στους μισθούς, να υπάρχει ανταγωνισμός σε όλα. Αυτό καθιστά την οικονομία ζωντανή η Βρετανική οικονομία παρά το Brexit ανθεί. Ενώ η ευρωπαϊκή οικονομία, η οικονομία του ευρώ δεν πάει και ιδιαίτερα καλά. Το ευρώ δεν πάει καλά. Οι γερμανικές τράπεζες έχουν προβλήματα, οι ιταλικές έχουν ήδη εξοκύλει. Κάθε προσπάθεια να βάλουμε όλα τα συστήματα της Ευρώπης σε ένα κουτί θα οδηγήσει σε κάτι, πώς να το πω, σοβιετικό κομμουνισμό, κάτι εξαιρετικά κακό και επικίνδυνο. Η Βρετανία δεν θέλει καμία σχέση με αυτό και αυτό είναι λόγος για να φύγουμε. Ακόμα ένας λόγος για να φύγουμε. Διαδικασία catch the eye, γκραπίνη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν καταλαβαίνω πολύ καλά τη θέση κάποιων συνάδελφων. Επικρατεί πλήρη σύγχυση ο στόχος δεν είναι ένα ενιαίο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Επουδενή. Απλά θέλουμε να σεβόμαστε τα δικαιώματα των διακινούμενων εργαζομένων. Θα πρέπει αυτοί που μετακινούν σε μια άλλη χώρα να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους ντόπιου εργαζόμενους. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε ελεύθερη κυκλοφορία χωρίς να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα αυτά των εργαζομένων. Πρέπει για παράδειγμα να δουλεύουν με τους ίδιους μισθούς με τους μισθούς των εργαζομένων που έχουν μόνιμη κατοικία σε αυτή τη χώρα. Η Αυστρία έχει μειώσει αυτές τις παροχές και ο πρωθυπουργός της Δανίας έχει ανακοινώσει ότι θα κάνει το ίδιο. Ε, θέλουμε μια ενιαία αγορά όμως, θέλουμε μια ενιαία Ευρώπη. Πώς θα γίνει. Δεν θα πρέπει να πληρώνονται με τον ίδιο τρόπο ε, αυτοί που προσφέρουν την ίδια εργασία. Ευχαριστώ. Κύριε Λένερ, θέλετε μπλε κάρτα για τον κύριο Κόμπορν. Να εξηγήσω όμω ότι στον κύριο Κόμπορν ότι αυτό πήρε από τον αρχικό χρόνο ομιλία από τι ομάδε. Θα σα δώσω το λόγο μετά τον επόμενο μιλητή. Ο κύριο Μαριά είναι πρώτο και μετά θα έχετε εσεί το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε τα ασφαλιστικά συστήματα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. δεύτερον η ευελιξία στην εργασία η οποία εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια και ιδίως το σύστημα των αποσπασμένων υπαλλήλων ένα σύστημα που δημιουργεί κοινωνικό ντάμπινγκ είναι αυτό που έχει περιπλέξει όλα τα ζητήματα. κανένα ασφαλιστικό σύστημα δεν θα πρέπει να μετατρέπεται σε σύστημα επιδότησης γειτονικών χωρών όπως έχει γίνει αυτή τη στιγμή με το ελληνικό σύστημα ασφάλισης έναντι των διακοσίων εργαζομένων στην ελλάδα από τη βουλγαρία. τρίτον καμία διάκριση σε όσους εργάζονται νόμιμα στα κράτη μέλη ταυτόχρονα όμως όχι πολιτική εξαγωγής επιδομάτων. το επίδομα ανεργίας στηρίζει όσους βρίσκονται σε ανεργία για να βρουν δουλειά επομένως θα τους στηρίζει όσο παραμένουν στη συγκεκριμένη χώρα. η μόνη δυνατότητα εξαγωγής θα πρέπει να αφορά τη σύνταξη εκεί είναι ένα δικαίωμα το οποίο κανείς μπορεί να κουβαλήσει και στη χώρα του. επομένως θα πρέπει να δούμε όλα τα θέματα αυτά όπως και το brain drain το οποίο έχει οδηγήσει σε αφέμαξη κοινωνικής ασφάλισης και Κύριε Λέναρτσε, ένα λεπτό έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν ήταν μπλε κάρτα, ήταν μάλλον διαδικαστικό το θέμα. Προφανώ ο κύριο Κόμπορν και οποιοδήποτε από το EFD δεν ε, ενοχλήθηκε να έρθει στην αρχή τη κάθε τέτοια συζήτηση και νομίζω ότι είναι λίγο άδικο μετά το πρωινό, το, τον υπνάκι του να εμφανίζεται εδώ και να του δίνουμε παρόλα αυτά χρόνο ομιλία. Αν πραγματικά μα νοιάζει η κάθε ομιλία, να έρχεται στην ώρα του ο καθένα. Αν δεν έρχεται στην ώρα του, μετά είναι δικό του το φταίξιμο. I'm a very fair Είμαι πολιτική πρόεδρο, λέει πρόεδρο, και νομίζω ότι αν κάποιο είναι στον κατάλογο ομιλητών ε, συνήθω του επιτρέπουμε να πάρουν το λόγο ακόμα και εκ των υστέρων αλλά το σημειώνουμε εν πάση περιπτώσει το θέμα σα για την επόμενη τέτοια ομιλία και συζήτηση που θα γίνει πρωί-πρωί. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μιλάντα. Με ανισχύει πολύ αυτή η συζήτηση. Ο σεβασμό των κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων για να αποφύγουμε την απάτη, τον αθέμητο ανταγωνισμό και την ανασφάλεια δικαίου μας, ε, μας κινητοποιεί. Για παράδειγμα, ε, για μας η κινητικότητα είναι η μετανάστευση στη Γαλλικία. Ε, έχουμε πάρα πολλούς που έχουν πάει στην Νορβηγία και ακόμα δεν έχουν λάβει παροχές ανεργίας κλπ στον... οι, Γαλλικοί, οι Γαλλικιανοί, οι οποίοι μετακινούνται στην Βόρεια Πορτογαλία, έχουν, αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Επίσης, κάποιοι που έχουν ε, μεταναστεύσει στη Σουηδία και γυρίζουν στη χώρα μας ε, δεν μπορούν να αναγνωρίσουν ε, την, την περίοδο κοινωνικής ασφάλισης εκεί πέρα. Εγώ έχω κάνει πολλές, ε, πολλά ερωτήματα, κοινωνιστικέ ερωτήσεις κλπ. για αυτά τα θέματα. Πρέπει να εργαστούμε έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την ίση μεταχείριση. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πιμέντε Αυτή η πρόταση που κάποιοι προσπαθούν να μπλοκάρουν ε, αποτελεί μεγάλη πρόοδο σε σχέση με την πρόταση της ε, Κομισιόν. Αλλά α είμαστε σαφεί. Ο συντονισμό των συστημάτων κοινωνική ασφάλισης μπορεί να γίνει μόνο αν υπάρχουν αυτά τα κοινωνικά, συστήματα κοινωνική ασφάλιση και είναι ανοιχτά, αλληλέγγυα και για όλου. Ε, αν αναδιανέμουν και εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Πριν από δύο εβδομάδες αναγνωρίσαμε, ε, υιοθετήσαμε ένα ε, ευρωπαϊκό σύστημα συντάξεων που οδηγεί, θα οδηγήσει στην ιδιωτικοποίηση του συστημάτου κοινωνική ασφάλιση. Ε, ε οι τελευταίες, ε, οι τελευταίες πρόοδοι που έγιναν στην Πορτογαλία με συνεισφορά μας είναι ανεπαρκής αλλά αποδεικνύουν ότι η αύξηση των μισθών και η στήριξη των συστημάτων κοινωνική ασφάλιση εξασφαλίζει τη βιωσιμότητά του και προφανώ τα δικαιώματα, κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται ο κατάλογο των αγωγητών. Η κυρία Τίσεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα και ζωντανή συζήτηση για το πολύ σημαντικό αυτό θέμα. Προτείναμε να εξυγχρονίσουμε τους κανόνες συντονισμού κοινωνικής ασφάλισης πριν από δυόμιση χρόνια. Έγκαιρα, λοιπόν. Και προτείναμε αυτή τη νέα πρόταση γιατί πρέπει να διαφυράξουμε την κοινωνική προστασία ενός αυξανόμενου αριθμού κινούμενων εργαζομένων. Εν ώψη των μεγάλων δημογραφικών αλλαγών στην Ευρώπη πρέπει να προσαρμόσουμε τους κανόνες για να προστατεύσουμε σωστά τα δικαιώματα των πολιτών. Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων υπάρχει μόνο αν οι μετακινούμενοι ε, εργαζόμενοι ε, διαφυλάσσουν την κοινωνική τους προστασία. Ο εξυγχρονισμός θα παράσχει στις εθνικές διοικήσεις καλύτερη εργαλεία για να ε, αντιμετωπίσουν την απάτη και τις καταχρήσεις θα υπάρξει καλύτερη λειτουργία των προϋθεσμιών μεταξύ των, των Εθνικών Αρχών Κοινωνικής Ασφάλισης. Να τονίσω επίσης την ασφάλεια δικαίου που παρέχεται στους εργαζόμενους, στις επιχειρήσεις ε, που, ε, και που ασκούν την, το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία. Αυτό είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε τον εξυγχρονισμό του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Ζητούμε λοιπόν από το Κοινοβούλιο ως Επιτροπή να υιοθετήσει την θέση αυτή σε πρώτη ανάγνωση, δείχνοντας έτσι στους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους ότι ενδιαφερόμαστε για τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης και ενδιαφερόμαστε για την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Διότι ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης είναι κρίσιμος για την ελεύθερη κυκλοφορία και ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων και των επιχειρήσεων είναι κρίσιμη για την εσωτερική αγορά. Έχω εμπιστοσύνη ότι το Κοινοβούλιο μέχρι και την τελευταία μέρα της θητείας του θα δείξει στους πολίτες ότι τα δικαιώματά τους μετράνε, ότι το Κοινοβούλιο θα δείξει στις επιχειρήσεις της Ευρώπης ότι κατανοεί τις ανάγκες τους, όπως και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και θα δείξει σε όλους ότι η Ευρώπη μπορεί να δώσει αποτελέσματα. Επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε να χρησιμοποιήσω ένα λεπτό από το χρόνο σας για να πω το εξή. Αυτή είναι η τελευταία μου παρέμβαση σε μια συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η συνεργασία μεταξύ Επιτροπής και ευρωβουλευτών, ιδίω τη Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, ήταν πάντα εξαιρετική. Νομίζω ότι πετύχαμε πολλά μαζί και θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τις επιτυχίες που καταφέραμε μαζί. Ευχαριστώ και ό,τι καλύτερο σε όλους σας. Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστούμε την κυρία Τάισον και είμαι βέβαιη ότι οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Απασχόλωση σα γνωρίζουν καλύτερα από ότι εγώ, αλλά θα ήθελα και εγώ προσωπικά να σα ευχαριστήσω για τη συνεργασία, για την... Ε, το γεγονό ότι πάντα είχατε κατά νου το συμφέρον του Ευρωπαίου πολίτη. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ και σα εύχομαι κάθε επιτυχία και στη μελλοντική σα σταδιοδρομία. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο για δύο λεπτά στον συγκεκριτή μα, τον κύριο Μπάλλα. Δύο λόγια μόνο. Ε, και εμένα είναι η τελευταία μου παρέμβαση. Ε, εγώ είναι, υποστηρίζω ότι υπάρχει υπόλωση μεταξύ αριστερά και δεξιά, αλλά μερικέ ε, φορέ κάποιοι που είναι προ τα δεξιά ίσω είναι πιο προοδευτικοί από κάποιου που είναι στα αριστερά. Ο Γκάντι έλεγε ότι πιστεύουμε ότι ο, το μίσο είναι ο εχθρό, αλλά στην πραγματικότητα ο εχθρό είναι ο φόβο. Και, έχω και άκουσα πολύ φόβο στα λόγια σήμερα, στι παρεμβάσει σήμερα το πρωί. Ε, και πολλοί μάλιστα λένε ό,τι να είναι. Ε, έξι μήνες περίοδος εξαγωγής έξι μηνών ε, μετά από 20 χρόνια εργασίας ε, θα είναι δήθεν κάποιο δώρο στους εργαζόμενους από την Ανατολή από τις ανατολικές χώρες. Όταν ξέρουμε όμως ότι το Κοινοβούλιο έχει δείξει ότι με αυτή την περίοδο έξι μηνών ε, τους δίνεται η δυνατότητα να ενταχθούν καλύτερα στην τοπική αγορά εργασίας από την περίοδο τριών μηνών. Ακούω από την άλλη μεριά κάποιου ε, κάποιους από, τη, βόρειες και δυτικές χώρες της Ευρώπης να μην λένε τίποτα για τις μεγάλες επιχειρήσεις που αυτές οργανώνουν το κοινωνικό ντάμπινγκ. Δεν είναι οι εργαζόμενοι των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, είναι οι επιχειρήσεις της Δύσης και του Βορρά της Ευρώπης. Και ποτέ δεν ζητάτε μέτρα για αυτές τις επιχειρήσεις προκειμένου να εξασφαλίσουμε ε, αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων. Βλέπω λοιπόν ότι σας εμπνέει ο φόβος. Ο φόβος αυτών των πολυεθνικών επιχειρήσεων τις οποίες δεν θέλετε να αντιμετωπίσετε. Και αυτό με λυπεί πολύ. πολύ. Γιατί πολλοί μιλούν για τη χώρα τους μόνο και όχι για το σύνολο των Ευρωπαίων εργαζομένων. Και ακόμα και κάποια ε, μειοψηφίε της ε, αριστεράς ε, μιλούν μόνο για τη χώρα τους. Γιατί, Γιατί προφανώς έρχονται, έρχονται οι ευρωπαϊκές εκλογές. Οπότε προσπαθούν να μιλούν μόνο για τους εργαζόμενου εργαζόμενους και όχι για τους εργαζόμενους όλης Ευρώπης και για τις επιχειρήσεις οι οποίες ε, θέτουν σε σύγκρουση τους μεν με τους δε. Κάνω μια έκκληση σε όλους τους προοδευτικούς αυτού του Ευρωκοινοβουλίου, σε όλους αυτούς που πιστεύουν πως η Ευρώπη έχει νόημα μόνο αν εξασφαλίζει πρόοδο για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως της εθνικότητάς τους. Αυτό είναι που κάνει την Ευρώπη Ευρώπη. Το κείμενο προφανώ δεν είναι τέλειο, δεν λύνει όλα τα προβλήματα, αλλά είναι ένα μήνυμα ενότητας και προόδου σήμερα, ένα μήνυμα ειρηνικών σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων για να πολεμήσουμε τον αθέμητο ανταγωνισμό που κάποιοι θέλουν να σπείρουν μεταξύ, ε, μεταξύ τους. Ευχαριστώ. Thank you to our... Ευχαριστούμε τον εισηγητή μα και μακάρι να μπορούσαμε να αντικαταστήσουμε το φόβο με την ελπίδα. Και επειδή έχω χρόνο και είμαι και σε διάθεση θα επαναλάβω έναν ποιητή Ιρλανδό, τον κύριο Χίνη, σε ό,τι αφορά την ελπίδα και την εκδίκηση. Απαγγέλει ένα ποίημα η πρόεδρος. Και με τις ε, κουβέντε αυτέ. Θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα πρωτού ξεκινήσει η επόμενη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Ελπίζω να περιλαμβάνει πολύ ελπίδα με τον Πρωθυπουργό της Λετωνία, τον κύριο Κάρεν. ευχαριστώ πολύ.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 Ξεκινάμε αμέσως διότι έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον παλιό συνάδελφο και τον ευχαριστούμε που δέχθηκε την πρόσκλησή μας να μιλήσει για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρεις πολύ καλά το κοινοβούλιο, ξέρετε πολύ καλά το, το κοινοβούλιο σήμερα, σπίτι σας είστε, έχουμε πολλά ζητήματα. Ξέρετε πολύ καλά τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη σημασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γνωρίζετε τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ που ήρθατε, όπως γνωρίζετε. Εμείς θέλουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι στο κέντρο των πολιτικών συζητήσεων για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης είσαστε ένα επίτιμο μέλος το ποντινά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μετά τη, αυτό το καλωσόρισμα σας δίνω απευθείας τον λόγο και ευχαριστώ εκ νέου για την παρουσία σας εδώ. Ε, ε, Άρχεται η ηλεκτρονική διαδικασία για το Catch the Eye μετά τις παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού κ. Κάριντς. augsti godātais tajani kungs juncker kungs Κύριε Πρόεδρε Ταγιάννη, κύριε Πρόεδρε Γιούνκερ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι φίλοι. Καταρχήν, χαίρομαι ιδιαίτερα που σας μιλώ για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, το μέλλον της Ευρώπης. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, για δέκα χρόνια περίπου, εργάστηκα, ήμουν στο Κοινοβούλιο, ως μέλος του Κοινοβουλίου και κατάφερα να μάθω κάποια πράγματα κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Όταν θέλουμε εδώ να απευθύνουμε μία, μία ομιλία, θα πρέπει τουλάχιστον τρεις γλώσσες να χρησιμοποιούμε, γιατί δάλλως δεν βγαίνει. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα θα μιλήσω και γερμανικά και γαλλικά. Τα γαλλικά με δυσκολεύουν βέβαια, γιατί καταλαβαίνω τη γλώσσα, αλλά για να απευθύνω ομιλία στα γαλλικά ζουρίζομαι. Θα συνεχίσω λοιπόν στα αγγλικά. Και γιατί είναι η τέταρτη γλώσσα μάλιστα. Μιλάμε για μια αλλαγή. Το τέλος της θητείας, οι επερχόμενε εκλογέ αποτελούν πραγματικά μια περίοδο περισυλλογή. Προτού όμω ε, κοιτάξουμε στο μέλλον, θέλω να κάνουμε και μια ιστορική αναδρομή για να το θέσουμε όλα αυτά στο σωστό πλαίσιο. Λετωνία, λοιπόν. Ευρώπη. Τι ενώνει τους Ευρωπαίους. Η κοινή ιστορία από την αρχαία Ελλάδα, την αρχαία Ρώμη, μέσω του χριστιανισμού που διαδόθηκε σε όλη την Ευρώπη και ο χριστιανισμός και ο πολιτισμός διαδόθηκε σε όλη την Ευρώπη και τελικά τα τελευταία προπήργια ήταν οι βαλτικές χώρες οι οποίες ακόμα δεν είχαν προσαρτηθεί σε αυτόν τον κοινό χώρο, τον πολιτισμικό και θρησκευτικό σε ό,τι αφορά την πολιτιστική και την θρησκευτική αυτή κληρονομιά μόλις στην 13ο αιώνα ο Παπάς είπε ναι σε μία σταυροφορία στις βαλτικές χώρες για τους μη χριστιανούς. Και έκτοτε η χώρα μας πέρασε όλες τις ε, πολιτισμικές εξελίξεις ε, και αναστατώσεις ε, που πέρασε και η υπόλοιπη Ευρώπη, τη μεταρρύθμιση, την αναγέννηση, ε, τον διαφωτισμό. Σήμερα η χώρα μας είναι λουθερανική κατά μεγαλύτερο βαθμό στο νότο και το ανατολικό κομμάτι πιο πολύ. Και θεωρούμε τον εαυτό μας μέσω της ιστορίας μας ήμασταν τμήμα του βορειοευρωπαϊκού πολιτισμικού χώρου και αυτό το λέμε με ρεαλιστικό τρόπο. Είμαστε ρεαλιστές, υπομονετικοί και θέλουμε να είμαστε πάντα μετριοπαθείς. Έχουμε μεγάλη δημιουργικότητα, μεγάλη επιχειρηματικότητα. Αυτό πάντα μας διέκρινε για εκατοντάδες χρόνια μετά την εισαγωγή και την... το χριστιανισμό στη χώρα μας. Αντιμετωπίσαμε διάφορες πολιτικές και στρατιωτικές αναστατώσεις από την Γερμανία, από την Πολωνία ενίοτε, από τη Σουηδία και άλλες φορές από τη Ρωσία. Σε όλη αυτή την φάση διατηρήσαμε την ταυτότητά μας και τη γλώσσα μας βέβαια. Και μόλις στα τέλη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου 1918 διακηρύξαμε την ανεξαρτησία μας επιτέλους. Πήρε άλλα δύο χρόνια ο πόλεμος της ανεξαρτησίας ε, να απελευθερώσει την χώρα από τα στρατεύματα τα γερμανικά και τα ρωσικά που ήταν στην ε, χώρα μας. Και ο παππούς μου, σε ό,τι αφορά την προσωπική μου ιστορία, μπήκε στον τσαρικό στρατό ως στρατιώτης ε, του Τσάρου και έγινε μετά πολσεβίκο στρατιώτης κατά της του Τσάρου και όταν άκουσε ότι η χώρα μα ανακήρυξε την εξαρτησία τη, έγινε πολεμιστή τη ελευθερία, υπέρ τη ανεξαρτησία. και αυτό αποτελεί ένα κλασικό παράδειγμα τη εποχή. Η χώρα μας αναπτύχθηκε λοιπόν μεταξύ των πολέμων στο Μεσοπόλεμο και μετά ήρθε και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Σε μεγάλες ζημιές προκλήθηκαν στην Ευρώπη και εδώ μπήκα και εγώ στην ε, εικόνα αυτή. Εγώ είμαι γιος μεταναστών του πολέμου το 1944 οι γονεί μου ήταν 18 και 14. Έφυγαν από τη Λετωνία στη Σουηδία. 55.000 περίπου Λετωνοί έφυγαν στη Σουηδία και κάποιοι πιο λίγοι στη Γερμανία όταν ο Σοβιετικό στρατός ερχόταν για δεύτερη φορά να καταστρέψει τη χώρα. Οι γονεί μου λοιπόν μεγάλωσαν στη Σουηδία, γνωρίστηκαν, παντρεύτηκαν και μετανάστευσαν στη ΣΥΠΑ όπου γεννήθηκα και εγώ μαζί με τις δύο αδερφές μου. Πρώτα ήρθα, μάλλον και πρώτη φορά στη Λετωνία το 1984. Τότε ήμουν ε, μαθητής στο Λύκειο, στο τελευταίο σχολείο μεταναστών στη Γερμανία για Λετωνού. Τότε για πρώτη φορά πήγα στη Λετωνία και ο κόσμο τότε ήταν διαφορετικό. Η χώρα ήταν διαφορετική, όλα ήταν γκρίζα. Ο κόσμο δεν γελούσε, δεν χαμογελούσε στον δρόμο. Σοβιετικοί στρατιώτε παντού. Όλα στα ρωσικά υπήρχε πραγματικά έλλειψη επενδύσεων σε οποιαδήποτε υποδομή, κτίρια, δρόμους, ε, γέφυρες. Πραγματικά αποσύνθεση επικρατούσε. Και όταν ξεκίνησε η αλληλεγγύη στο τέλος του, της δεκαετίας του 80 και έπεσε και το τείχος του Μερολίνου στο 89, ξεκίνησε η αλλαγή. Το 91 επιτέλους ε, αποκτήσαμε την εξαρτησία μας και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αναπτύξαμε δημοκρατικούς θεσμούς. Αναπτύξαμε ελευθερή επιχειρηματικότητα, τραπεζικό σύστημα, οικονομία της αγοράς, από το τίποτα, από το μηδέν. Το 2004, 13 μόλις χρόνια μετά την ανεξαρτησία μας, μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Μέσα σε λίγες εβδομάδες θα γιορτάσουμε τα 15 χρόνια από την προσχώρησή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορώ να σας πω εξ ονόματος της χώρας μου ολόκληρη ότι δεν έχουμε μετανασ... μετανιώσει την προσχώρησή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε μία ημέρα. So what, what is, what is the EU? Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση? Πρώτα πρώτα, και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε, είναι μια ένωση αξιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου ιστορικά στην Ευρώπη. Πώς λύνονταν οι διαφορές. Με όπλα, με στρατιώτες, με τάγκς, με καταστροφή. Σήμερα πώς λύνουμε τις διαφορές. Με κουραστικές συζητήσεις, ε, διαφωνίες, ψηφοφορίες, αλλά με τρόπο διαφορετικό από ό,τι γινόταν στο παρελθόν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και σαν στόχο την οικονομική ανάπτυξη και στο κέντρο της είναι η ενιαία αγορά. Ανοίγοντας τα σύνορά μας οι μεν στου δε, δημιουργήσαμε μία από τις μεγαλύτερες αγορές στον κόσμο. 500 εκατομμύρια άτομα που πάνω κάτω είναι αντίστοιχη αγορά με αυτή τον ΙΠΑ που θεωρείται η ισχυρότερη οικονομία. Τα πράγματα ωστόσο δεν είναι όλα καλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι γνωρίζουμε ως πολιτικοί ότι υπάρχει ισχυρό αντιευρωπαϊκό αίσθημα. Υπάρχουν πολιτικοί που παρέχουν απλουστευτικές απαντήσεις σε σύνθετα, πολύ σύνθετα ζητήματα. Τους χαρακτηρίζουμε γενικά ως λαϊκιστές. Με απλά μηνύματα, ε, το, το μήνυμά μου είναι μην ε, πολεμάτε τους λαϊκιστές, αλλά αντίθετα ακούστε γιατί ο κόσμος ακούει Προσπαθήστε να καταλάβετε γιατί ο κόσμος ακούει τους λαϊκιστές και είναι δυσαρεστημένος. Πηγαίνετε λίγα χρόνια πίσω, 2008-2009. Μία τράπεζα κατέρευσε στις Ηνωμένε Πολιτείε. Καταραίων που και που. Αυτό οδήγησε σε μια αλυσιδωτή αλλαγή τραπεζικών κρίσεων ανά τον κόσμο, ιδίω στην Ευρώπη, που οδήγησε σε μια οικονομική κρίση. Τη μεγαλύτερη μετά την κρίση του 1929. το ΑΕΠ τη χώρα μου έπεσε σχεδόν κατά το 1 τέταρτο και σε άλλες χώρες μειώθηκε το ΑΕΠ ίσως όχι τόσο πολύ. Βγαίνοντας από την οικονομική κρίση, τι συνέβη λίγα χρόνια μετά, η μεταναστευτική κρίση, η ανασφάλεια, η, η, η πόλεμη στην Μέση Ανατολή οδήγησε σε μετακινήσεις πλεισμών, πρόσφυγες και μετανάστες. Αποτέλεσμα είναι αυτό που εγώ χαρακτηρίζω ως πολιτική κρίση. Ο κόσμος χάνει την εμπιστοσύνη του στο σύστημα. Είναι κατανοητό αυτό. Πρέπει να τους βοηθήσουμε να ξανααποκτήσουν την εμπιστοσύνη τους. Αν δείτε τους ε, ψηφοφόρους, θα δει ποιες είναι οι βασικές τους ανησυχίες. Τέσσερις θα έλεγα. Δουλειές, τρόπος ζωής, μετανάστευση, περιβάλλον και ασφάλεια. Για να μιλήσουμε για το μέλλον στην Ευρώπη πρέπει να μιλήσουμε για τα τέσσερα αυτά θέματα. Δουλειές πρώτα-πρώτα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έναν μηχανισμό για ταχύτερη ανάπτυξη των θέσεων εργασίας. Αυτό που αποκαλούμε ενιαία αγορά. Θυμάμαι μια ιστορία όταν ήμουν παιδί. Μπορεί να είναι ένας μύθος του εσώπου, δεν ξέρω. Ένα παιδί, είχε, ένας πατέρας είχε τρία παιδιά. Δίνει ένα μπαστούνι στον ένα και του λέει σπάστο. Και το παιδί το σπάει. Το δίνει στο δεύτερο και το δεύτερο και του λέει σπάστο. Το σπάει και αυτό. Και στον τρίτο του δίνει ένα πακέτο με, μπαστού, με, με, με μπαστούνια και του λέει σπάστα και αυτός δεν μπορεί να τα σπάσει. Το, το, το, αποτέλεσμα, το, το, το ηθικό δίδαγμα από αυτό είναι ότι όταν είσαι μόνος σου σπάς εύκολα, όταν είσαι ενωμένο, είσαι ισχυρός. Και αυτό είναι το θετικό της ενίας αγοράς. Έχουμε μια σειρά προκλήσεων για την ενία αγορά απ' έξω η άνοδος της Κίνας. Η, μια κυβέρνηση τον ΗΠΑ που δεν πιστεύει τόσο πολύ ότι μπορεί να παίξει πλέον ένα μείζωνα ρόλο στην παγκόσμια οικονομία και στο παγκόσμιο εμπόριο. Κίνα πρώτα. Είναι μια χώρα που ανοιχτά επιδοτεί τις τεράστιες βιομηχανίες της, οι οποίες έρχονται στην Ευρώπη και ανταγωνίζονται χω, άνισα με ε, συγκριτικό πλεονέκτημα. Τι απαντάμε εδώ. Η απάντηση στον αθέμητο ανταγωνισμό, λέω, δεν είναι ο προστατευτισμός. Δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τον δρόμο των Κινέζων. Δεν θα πρέπει να γίνουμε σαν τους Κινέζους, να ζητήσουμε από τους Κινέζους να γίνουν σαν και εμάς, ανοίγοντας την αγορά τους. Έχουμε πολύ ισχύ ως Ένωση και ως ενία αγορά. Αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Όχι σαν μικρά μπαστούνάκια, αλλά σαν ένα, ένας βεσμός από ε, κράτη που μπορούν να επηρεάσουν τον κόσμο. Τώρα, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε κάποια εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσουμε, που σχετίζονται με τα εσωτερικά εμπόδια στην ενιαία αγορά. Ιδίως στην ψηφιακή σφαίρα και στις υπηρεσίες αναρωτηθείτε όπως αναρωτιέμαι και εγώ. Γιατί οι μεγαλύτερες εταιρείες του ίντερνετ προέρχονται από τις Ηνωμένε Πολιτείε και δεν είναι ευρωπαϊκές. Η απάντηση είναι προφανής. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχει μια ζώνη δολαρίου, μια ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ομοσπονδιακό προπολογισμό και μηδενικά εμπόδια μεταξύ των πολιτιών στο εμπόριο. Έχουν μια πραγματικά ενωμένη ενιαία αγορά, μικρότερη από εμά, 330 εκατομμύρια κατοίκου. Έχουμε μεγαλύτερη αλλά πολλά εμπόδια. Όταν λοιπόν λέμε ότι θέλουμε να έχουμε εθνικούς πρωταθλητές, δεν θα πρέπει να κάμπτουμε την ε, νομοθεσία για τον ανταγωνισμό για να δημιουργούμε τεχνητά εθνικούς ε, πρωταθλητές, αλλά να μειώνουμε τα εμπόδια στο εσωτερικό της αγοράς για να αναπτυχθούν πραγματικά αυτοί οι πρωταθλητές και να ανταγωνιστούν τις ΗΠΑ και την Κίνα. Ένας από τους ακρογωνιαίους λήθους της ενίας αγοράς είναι το χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι τράπεζες. Πριν από 10 χρόνια η μεγαλύτερη απειλή εναντίον αυτών ήταν η ρευστότητα. Οπότε δημιουργήσαμε την Τραπεζική Ένωση έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Εντοκή Τράπεζα να επιτηρεί ε, τις πιο μεγάλες από αυτές. Από τότε όμως ο κόσμος έχει αλλάξει. Η ρευστότητα δεν είναι πλέον το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ένα νέο πρόβλημα προέκυψε που είναι η τρομοκρατία και η χρηματοδότηση τρομοκρατία στην Ευρώπη. Και πώ συμβαίνει αυτό πολύ συχνά μέσω παράνομων μεταφορών μέσω του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματος. Οπότε πού είναι η νομοθεσία μας για το ξέπλυμα χρήματο. Με την κυρία Σαρτζεντίνη ήμουνα συνεισηγητής παλιότερα για αυτό το θέμα και έμαθα αρκετά πράγματα. Η νομοθεσία κατά του ξεπλήματος ε, χρήματος έχει σχέση, ε, άμεση σχέση με την αξιολόγηση κινδύνου και με την αποφυγή του βρώμικου, χρήματος να μπαίνει, ε, να, βρώμικο χρήμα να μπαίνει στο τραπεζικό μας σύστημα. Για τα τελευταία 20 χρόνια ποσά από την Ρωσία προσπαθούν να βγουν από τη Ρωσία. Γιατί, Γιατί η Ευρώπη είναι ασφαλής, έχει ασφάλεια δικαίου, κράτος δικαίου και κανείς δεν σου αρπάζει τα χρήματα ε, πολλά από αυτά τα χρήματα που έρχονται από τη Ρωσία είναι καθαρά, αλλά κάποια όχι. Αυτοί οι εγκληματίε που προσπαθούν να φέρουν χρήματα από τη Ρωσία στην Ευρώπη, δεν μιλώ για αυτού που προσπαθούν να ε, βελτιστοποιήσουν ε, το φόρο πληρών κλπ. Μιλώ για ανθρώπου οι οποίοι ε, θέλουν να φέρουν βρώμικο χρήμα. Αυτοί, σαν γεράκια, υπερίπτανται και προσπαθούν να βρουν του αδύναμου κρίκου στην αλυσίδα. Εδώ σε αυτή τη χώρα μπορεί να κάνει αυτό, σε εκείνη τη χώρα μπορεί να, δεις κάτι άλλο, να κάνει κάτι άλλο κλπ. Ε, και εμεί ήμασταν τμήμα αυτή τη αλυσίδα. Ε, το, όμως δεν είμαστε μόνοι μας, ε, το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό. Από τότε που έγινα πρωθυπουργό, δεν μπορώ να περιμένω όλοι να συμφωνήσουμε, οπότε εγώ καθαρίζω το σπίτι μου. Θα έχουμε το πιο καθαρό και ανθεκτικό τραπεζικό σύστημα στην Ευρώπη. Σε 1,5 χρόνο θα μπορούμε να σα ενημερώσουμε τον καθένα σα ε, ξεχωριστά και όλου μαζί για το πώ μπορεί να καθαρίσει κανεί το τραπεζικό σύστημα. Θα διώξω τα ποντίκια από το δικό μου σπίτι. Και το δικό μου σπίτι θα είναι καθαρό. Αλλά τι θα γίνει με του γείτονε. Οι εγκληματίε μπορεί να εγκατέλειψαν τη Λετωνία, αλλά είμαι σίγουρο πω δεν εγκατέλειψαν την Ευρώπη. Οπότε θα πρέπει να ε, καθαρίσουμε όλη τη γειτονιά. Αυτό σημαίνει ότι η τραπεζική εποπτεία για την καταπολέμηση του, ε, του, του ξεπλήματος θα πρέπει να είναι βασική μας μέρημνα. Ε, μια άλλη, ανησυχία των ψηφοφόρων είναι το, το τρόπο ζωή του και η μετανάστευση. Εδώ δεν υπάρχουν απλές απαντήσεις, δεν έχω εγώ απλές απαντήσεις και δεν νομίζω ότι κανεί έχει. Η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη είναι ένας εξαιρετικό προορισμό για να ζήσει κανεί και να εργαστεί. Σταθερέ οικονομίε, σταθερέ δημοκρατίε κράτος δικαίου, ε, ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες, ενώ πολλοί από τους γειτονές μας δεν έχουν κάτι τέτοιο. Οπότε η πίεση, οι πιέσεις, ε, μεταναστευτικές πιέσεις αυξάνονται. Και δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα εξαλειφθεί, θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Η χώρα μου δέχτηκε κάποια μετανάστευση. Πάνω από 700.000 άτομα μετανάστευση έφτασαν στη χώρα μου κατά τη διάρκεια του Σοβιετικού καθεστώτος. Το 1 τρίτο του πληθυσμού μας. Έτσι είμαστε 2 εκατομμύρια. Δεν είχαμε κυβέρνηση τότε, οπότε <laughs> δεν πήραμε εμεί αυτέ τι αποφάσει. Τι αποφάσει λαμβανόντουσαν από τη Μόσχα. Δεν υπήρχε διαδικασία συναπόφαση, δεν είχαμε λόγο. Με, αφού ανεξαρτοποιήθηκαμε, πώ το αντιμετωπίσαμε μέσω της ένταξης. Αυτή είναι η λέξη κλειδί. Πρέπει να συνεργαστούμε με αυτούς, με το, να προσαρμόσουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα έτσι ώστε αυτοί οι μετανάστες να ενταχθούν στη δική μας κουλτούρα. Αυτό είναι ο, ο μόνος τρόπος. Ε, δεν μπορεί κανείς να το αποφύγει αυτό. Δεν μπορεί κανείς να αποφύγει ότι κάποιοι θα θέλουν να έρχονται συνεχώς στην Ευρώπη. Θα πρέπει να τους εντάσσουμε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε για να μετριάσουμε τις ροές είναι τα εξωτερικά σύνορα, η Frontex. Είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα που πρέπει να ενισχυθεί. Αν αποδείξουμε στους ψηφοφόρους μας ότι ελέγχουμε τα εξωτερικά μας σύνορα, μπορούμε να έχουμε ελεύθερα εσωτερικά σύνορα. Θυμάστε πόσο εύκολο ήταν παλιότερα ε, να κυκλοφορεί κανείς στη ζώνη του Σέγγεν. Ε, μεταξύ για παράδειγμα Στρασβούργου και Γερμανίας. Τώρα πια πολλές φορές οι γέφυρες κλείνουν, ξανά τοποθετούνται τα σύνορα. Ε, αυτό θα πρέπει να το αποφύγουμε. Αλλά γι' αυτό χρειαζόμαστε ισχυρά εξωτερικά σύνορα και χρειάζεται να χρηματοδοτήσουμε ε, ε, καταβλισμούς προσφύγων και μεταναστών. Χρειάζεται να συνεργαστούμε με τρίτες χώρες και να τις χρηματοδοτήσουμε και οπωσδήποτε θα πρέπει να εργαστούμε πάνω στην ένταξη των μεταναστών. Είμαστε μια ένωση 28 ακόμα κυρίαρχων κρατών, το καθένα με τη δική του εθνική ταυτότητα, οπότε είναι εξαιρετικό, εξαιρετικά σημαντικό να διατηρήσουμε την κουλτούρα μας, τη γλώσσα μας και την εθνική μας ταυτότητα. Αυτό μέσω της ένταξης, της ενσωμάτωσης όσων έρχονται στη χώρα μας, στις χώρες μας και θα πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτό θα πρέπει να εργαστούμε. Αν αποδείξουμε ότι ελέγχουμε τα εξωτερικά σύνορα και μπορούμε να εντάξουμε τους μετανάστες, οι ψηφοφόροι θα χαλαρώσουν σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Τρίτη ανησυχία τους, το περιβάλλον. Η κλιματική αλλαγή είναι αληθινή. Είναι κάτι το αληθινό ένα γεγονός. Ο άνθρακας και η... Ε, ορυκτοί υδρογονάνθρακες εξακολουθούν να καίγονται και επιβαρύνουν το περιβάλλον. Οπωσδήποτε θα πρέπει να πάρουμε πολλά μέτρα και επιλαμβάνουμε ε, ενεργειακή αποδοτικότητα κλπ. Το σημαντικό όμως είναι το ενεργειακό μείγμα. Εμείς είμαστε δεύτεροι μετά τη Σουηδία σε ό,τι αφορά τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, 45% του συνολικού μα μείγματο. Δεν είναι όλε οι χώρε έτσι. Πολλέ χώρε εξαρτώνται πολύ περισσότερο από τον άνθρακα. Δεν μπορούμε όμως να μειώσουμε του, τη χρήση του άνθρακα με επιθυμίες. Κάποιος πρέπει να πληρώσει αυτή τη μετάβαση και θα χρειαστεί χρόνος. Ανεξαρτητός όμως του πόσο γρήγορα μπορούμε να προχωρήσουμε, υπάρχει μία διαστατική αλλαγή που πρέπει να γίνει έτσι ώστε να επιταχυνθεί η μετάβαση. Και πάλι αυτό είναι το άνοιγμα της ε, αγορά ενέργεια στον ανταγωνισμό. Χρειάζεται ανταγωνισμό στι ανανεώσιμε. Για παράδειγμα, αγορά ηλεκτρική ενέργεια. Πολλέ χώρε ε, έχουν ρυθμίσει ε, το θέμα τη ενέργεια, τον, αγορα ώρα ενέργειας, οπότε οι καταναλωτέ πληρώνουν το ίδιο ανεξάρτητα από την ώρα τη ε, μέρα ή από τη μέρα τη εβδομάδα. Οπότε δεν σε νοιάζει. Μπορεί να βάλει το πλυντήριό σου να δουλέψει όποια στιγμή τη μέρα, όποια μέρα τη εβδομάδα θέλει. Όταν όμω ανοίγουμε τις αγορές μας στον ανταγωνισμό. Ή ο ανταγωνισμός ε, δίνει κίνητρα και αντικίνητρα με μειώσεις τιμών ή αυξήσει τιμών ανάλογα με την ώρα της μέρας, τη μέρα της εβδομάδας. Οπότε μειώνουμε ε, τις ε, ανάγκες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στις ώρες εχμής. Ε, Αν μπορούμε σε αυτέ τι ώρε αιχμή, για παράδειγμα, να επιτρέψουμε στα ψυγεία να αυξήσουν τη θερμοκρασία του κατά ένα-δύο βαθμού, αυτό μα εξοικονομεί πάρα πολύ ενέργεια. Για αυτά τα πράγματα χρειαζόμαστε ανταγωνισμό και χρειαζόμαστε απορρίθμιση. Τέταρτη ανησυχία των πολιτών μας η ασφάλεια. Αυτό σημαίνει κάτι διαφορετικό ε, για τον Νότο, διαφορετικό για τον Βορρά. Στο Νότο, όταν μιλάμε για ασφάλεια, ε, ε, το μυαλό πηγαίνει πιο πολύ στην ανεξέλεγκτη μετανάστευση και στην τρομοκρατία. Στη Δυτική Ευρώπη, η μεγαλύτερη απειλή εναντίον της ασφάλειας είναι το ανεξέλεγκτο Brexit ενδεχομένω και για το εμπόριο, αλλά και για την ειρήνη στην Βόρεια Ιρλανδία. Εγώ προέρχομαι από τη Λετωνία. Όταν εμείς έχουμε στο μυαλό μας την ε, μιλάμε για ασφάλεια, έχουμε στο μυαλό μας τη Ρωσία. Ε, αυτό είναι κοινό μυστικό. Ε, η Ρωσία είναι ένας γείτονας που έχει μια κυβέρνηση που έχει μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική. Πιστεύει ότι περικυκλώνεται από εχθρούς που είναι έτοιμοι να τις επιτεθούν. Αυτό είναι το <laughs> αμυντικό δόγμα της Ρωσίας. Ε, οπότε προσπαθεί να αποδυναμώσει τους γειτονές της. Αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη απειλή από τη Ρωσία δεν είναι στρατιωτική. Και το στρατιωτικό είναι απειλή, αλλά δεν είναι η μεγαλύτερη απειλή. Έχουμε το ΝΑΤΟ, έχουμε τη δική μας προετοιμασία. Η μεγαλύτερη απειλή είναι τα ψεύδη και οι ψεύτικες πληροφορίες ή ψευδείς πληροφορίες, fake news. Ζούμε στον κόσμο αυτών των πολυόμορφων συσκευών, όλοι έχουμε από μία τουλάχιστον Πίστευα, όπως όλοι μας παλιότερα, ότι θα μας εξασφαλίσουν αυτές οι συσκευέ απόλυτα ελεύθερη ε, πρόσβαση στις πληροφορίες. <laughs> Και γίνεται αυτό. Απ' την άλλη μεριά, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει ένας τρομακτικά καλός τρόπος για την διάδοση ε, χωρίς καμία καθυστέρηση ε, ψευδών ειδήσεων. Και όλο και περισσότερος ε, κόσμος εγκαταλείπει ε, τη, αξιόπιστα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τους υπεύθυνους δημοσιογράφους που ελέγχουν τις πληροφορίες κλπ. και πιστεύει ε, πέφτει θύμα ψευδών πληροφοριών που διαδίδονται μέσα στο διαδίκτυο. Οπότε έχουμε ευθύνη για τις πλατφόρμες που ε, διαδίδουν στο ίντερνετ αυτές τις πληροφορίες. Προφανώς είναι ολιστηρός ο δρόμος, γιατί είναι πολύ λεπτή η γραμμή ανάμεσα στην ε, ευθύνη ε, και ε, στη φήμωση, στη λογοκρισία. Δεν θα υποστηρίξω ποτέ τη λογοκρισία, αλλά θα πρέπει να βρούμε το όριο. Γιατί πρέπει να δούμε τι προσπαθούν να κάνουν. Προσπαθούν να διχάσουν την κοινωνία, να μας ε, φέρουν σε σύγκρουση μεταξύ μας. Για παράδειγμα, εμβολιασμοί. Από πού ξεκίνησε το επιχείρημα ότι οι εμβολιασμοί οδηγούν σε αυτισμό. Οι Ρώσοι ξεκίνησαν αυτή, αυτό τον ισχυρισμό. Και η, ε, η αποφυγή του εμβολιασμού δημιουργεί πολλά προβλήματα στην Ευρώπη. Μετανάστευση και στη μετανάστευση πολλά τα ψεύδι που ξεκινούν από τη Ρωσία, το Brexit. Έχει γίνει, ο Τζορτ Σόρος έχει γίνει μια φούσκα στην Ανατολική Ευρώπη ότι δήθεν ε, συνωμοτικά επηρεάζει τη ζωή όλων μας κλπ. Αν δεν δεχτούμε το, την πραγματικότητα δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Η, για την ασφάλεια ε, η στρατιωτική απειλή δεν είναι τόσο μεγάλη. Ε, Παρ' όλα αυτά, εμείς επενδύουμε 2% του προπολογισμού μας στην ασφάλεια και, και όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ πρέπει να κάνουν το ίδιο. Απ' την άλλη μεριά, εξίσου σημαντικό είναι να αντιμετωπίσουμε το θέμα των ψευδών ειδήσεων. Και εκεί μάλλον θα πρέπει να εξετάσουμε το κατά πόσο αυτό μπορεί να γίνει μέσω νομοθεσίας. Τέλος, ε, έχω και κάποια θέματα σχετικά με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο θέλω να, ε, τα οποία θέλω να σας σχολιάσω. Πρόκειται για τον 7 η προπολισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνο, όπως και εσείς, ότι θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερα στην έρευνα και τεχνολογία στην Ευρώπη. Έχουμε πολλούς νέους έξυπνους ευφύς ανθρώπους που θα πρέπει να τους κρατήσουμε στην Ευρώπη και να τους αναπτύξουμε εδώ. Όμως, εξίσου σημαντικό είναι αυτή η επένδυση να μην γίνεται μόνο σε ορισμένα σημεία της Ευρώπης, αλλά σε όλη την Ευρώπη. Γιατί έξυπνα μυαλά υπάρχουν παντού στην Ευρώπη. Όλη η Ευρώπη χρειάζεται επένδυση στην αριστεία. Η αριστεία δεν μπορεί να επικεντρωθεί μόνο σε 2, 3, 4, 5 πρωτεύουσε. Ναι, λοιπόν, στην έργα την ανάπτυξη, αλλά θα πρέπει να διαχυθεί σε όλη την Ευρώπη. Η ευφυή συνοχή. Η συνοχή εξακολουθεί να είναι ε, σημαντική, αλλά θα πρέπει να είναι ευφυή. Θα πρέπει οι πιο φτωχέ περιοχέ να συγκλίνουν προ τι πιο πλούσιε. Αυτό πρέπει να το διασφαλίσουμε. Τέλο, το θέμα των αγροτών στην Ευρώπη. Ο ευρωπαϊκό προπολογισμό παλιότερα αφιερωνόταν σε πολύ μεγάλο βαθμό στην ΚΑΠ. Όχι τόσο όσο παλιά, αλλά εξακολουθεί αυτό το φαινόμενο και σήμερα. Είναι ιστορική ευκαιρία μας να ε, εξαλείψουμε μια ιστορική αδικία. Αυτή τη στιγμή επιδοτούμε μέσω άμεσων πληρωμών τους γεωργούς μας. Υπάρχει όμως μια παγίδα. Οι επιδοτήσεις δεν είναι ισότιμες, παρόλο που τα προϊόντα τους διατίθενται με ισότιμους τρόπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί που είναι οι λιγότερο ευνοημένοι είναι οι βαλτικές χώρες. Για μαθηματικούς λόγους που σχετίζονται με τα δεκαετία του 90, εμείς επιδοτούμαστε λιγότερο σε σχέση με άλλους. Οι δικοί μας γεωργοί ανταγωνίζονται με ίσους όρους με τους υπόλοιπους γεωργούς, αλλά αυτό θα ήταν πραγματικά ισότιμο αν επιδοτούνται με τον ίδιο τρόπο. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται να μειώσουν, να χαμηλώσουν το βιωτικό τους επίπεδο για να μπορούν να ανταγωνίζονται με θεμητό τρόπο. Αν συνεχίσουμε την επιδότηση,